σαν προβλήματα. Το ψήφισμα που υπέβαλαν τα πολιτικά κόμματα είναι ένας καλός συμβιβασμός και θέλω να τον υποστηρίξω. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί για την ομάδα της Ευρώπης, της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας ο κ. Μπέλντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.